Συνάδελφοι, επαναλήψη της συνεδρίασης, επόμενο σημείο, έγκριση συστάσεων. Η γραμματεία διένυμε, διένυμε τον κατάλογο ψηφοφορία με τις τροπολογίες, οπότε για κάθε παράγραφο θα σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή όχι. Μία προς μία. Ακούστε με παρακαλώ προσεκτικά. Δεν έχουμε συζήτηση, μόνο ψηφοφορία. Πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 1. του κυρίου Βουλευτή. Υπάρχει συμβαστική τροπολογία εδώ. Σημείωσε τις ε, συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των πολιτών στο Μαυροβούνιο και καλεί τις κρατικές αρχές να διερευνήσουν το ταχύτερο δυνατόν με τρόπο αποτελεσματικό τις καταγγελίες περί διαφθοράς κλπ. Αυτό είναι η συμβαστική. Οπότε, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ποιος είναι υπέρ. Να, να, μια εξήγηση, επεξήγηση τροπολογίας της συμβαστικής. Παρακαλώ. Όχι, κοιτάξτε, όχι, όχι. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την τροπολογία. Το είχαμε πει και την περασμένη φορά. Συγγνώμη, πού, πού, πού το γράφει ότι δεν μπορούμε να επεξηγήσουμε την τροπολογία. Σε ποιο, ποιος το λέει αυτό. Όχι, απαγορεύεται η επεξήγηση. Όχι. Κύριε Κρυβοκάπιτς, ε, δεν έχετε δίκιο. Έχω προεδρεύσει πάνω πολλέ φορέ. Αυτό είναι ο κανόνα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαίωμα επεξήγηση. Το λέει και ο συμπρόεδρό μου. Τι είπα, ψηφίζουμε και μόνον. Πρέπει να εξηγήσω την ε, τροπολογία μου, λέει ο κύριο Κρυβοκάπιτς. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Εγώ θα επερμηθώ των δικών μου τροπολογιών, θα πρέπει να εξηγήσω. Ε, κάποιος να μιλήσει ένας υπέρ, ένας κατά. Ε, αυτό είναι το, το ελάχιστο, συγγνώμη. Αν δηλαδή κάποιος επιθυμεί να το πράξει, εννοείται ότι μπορεί. Είδατε, ε, θέλουν να σταματήσουν το μποϊκοτάρισμα. Ε, θέλουν να, να, να μας μποϊκοτάρουν τώρα με τη σειρά τους. Ε, αγαπητοί συναδελφοί, στι τρει τελευταίε συνεδριάσει δεν είχαμε επεξηγήσει. Είχαμε συμφωνήσει οι δύο συμπρόεδροι. Ήσασταν εδώ. Ήσασταν εδώ. Και έχω και πολλού μάρτυρε. Ήσασταν εδώ, κυρία. Εν πάση περιπτώσει, μόνο προτείνων έχει ένα λεπτό. Επειδή είναι συμβαστική να τη διαβάσω, μπορώ παρακαλώ. Να εξηγήσω τη δική μου, λέει ο κύριος Κρυβόκαπιτς, Όπω όπως έχετε δει στο σχέδιο, δεν υπήρχε καμία αναφορά στις διαμαρτυρίες, στις διαδηλώσεις. Ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το Μαυροβούνιο αυτή τη στιγμή. Οπότε, προτείνω μια συμβαστική. Βλέπω ότι εν μέρη αποδεχθήκατε την συμβαστική μας. Καλό αυτό. Θα ήταν χρήσιμο για το μέλλον, για όλους μας για εσάς. Τέλος πάντων, επιμένω επί της μου αλλά καλή και συμβαστική. Συναδελφοί, ρωτώ τον ε, συμπρόεδρο. προτείνω την συμβιβαστική. Οι δύο συμπρόεδροι προτείνουν την συμβιβαστική. Μα συγγνώμη, λέει ο κύριο Κρυβό Καπίτσο, δεν την έχουμε δει. Να, να τη δούμε. Δεν την έχω λάβει, δεν είμαι μόνο εγώ. Κανεί δεν έχει δει το κείμενο να τη δεχθούμε, αλλά να τη δούμε πρώτα. Θα σας τη διαβάσω αργά. Τι θέλετε να κάνουμε, λέει ο κ. Καπίτσο. Κοιτάξτε, στη Βουλή μας, ακόμα και στη δική μας Βουλή, δεν μπορείς να ψηφίσεις για κάτι που δεν έχεις δει. Μισό λεπτό, ακόμα και στην Ολομέλη με 751 βουλευτέ έχουμε και προφορικές τροπολογίες. Κατά την άποψή μου, κυρία Καπίτσου, μπορούμε να ψηφίσουμε λίμωνο. Ωραία, διαβάζω την συμβαστική τροπολογία και να ψηφίσουμε. Διαβάζω. Σημειώνει τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των πολιτών του Μαυροβουνίου. Καλεί τι κρατικέ αρχέ να διερευνήσουν το σημαντικό δυνατόν και αποτελεσματικά τι καταγγελίε περί διαφθορά και υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου είναι πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ποιος ε, είναι υπέρ από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρακαλώ πρώτα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Όχι. Πολύ ωραία. Και τώρα οι συναδελφοί από το Μαυροβούλιο. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Όχι. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται η συγκεκριμένη συμβαστική τροπολογία. Όχι, δεν ψηφίσουμε τη δική σας τροπολογία, κύριε Κρύβα Κοπέτσι. Τη συμβιβαστική. Εκτός να αλλάξει τη θέση του ο συμπρόεδρος. Όχι. Όχι. Ψηφίσουμε μόνο τη συμβιβαστική. Τελείωσε. Έτσι γίνεται σε αυτήν την μεικτή επιτροπή. Ε, από τη στιγμή που υπάρχει συμβαστική, ε, καταπίπτουν όλες οι άλλες. κρυβό Καπίτσο. Μισό λεπτό. Η συμβαστική δεν είναι της Επιτροπής, είναι του Προέδρου, εν προκειμένου ή των συμπροέδρων. Εγώ έχω δικαίωμα να θέσω ψηφορία τη δική μου τροπολογία. Συγγνώμη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ε, υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία η συμβαστική, τελειώσαμε. Εκτός αν καταπέσει, αλλά αυτό δεν συνέβη σήμερα. Πάμε στην 2. Τροπολογία 2 του κυρίου Κρυβό Καπίτσου. Έχετε ένα λεπτό κύριε Κρυβό Καπίτσου, αν θέλετε να εξηγήσετε. Να τονίσω τι γίνεται με τα δικαιώματα των ανθρώπων στην κρατική τηλεόραση και με τον ε, διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ μιλάμε για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και αλλοιώθηκε η βούληση της η λειτουργία της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο κάπτει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και φανείς πρακτικές, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Και τονίζουμε εδώ ε, αυτά τα κοινοφανή χαρακτηριστικά του συστήματος στο Μαυροβούνιο αυτά. Ελπίζω να μην έφτασε το λεπτό. Με συγχωρείτε, δεν είναι καινούργια στοιχεία αυτά. Μιλάμε για δικαστικές αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται. Αλλά μιλήστε με το ανώτατο δικαστήριο. Τα τακτικά δικαστήρια δεν μπορούν να αποφανθούν για τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Εν πάση περιπτώσει ψηφίζουμε τώρα την ε, τροπολογία 2 του κυρίου Κρυβόκαπιτς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτα. Ποιο είναι υπέρ. Τρία. Ένα. Και τώρα. Από το Μαυροβούνιο. Υπέρ. Κατά. Οχτώ. Αποχή. Άρα οι δύο Απορρίπτεται. Τρία. Το πρώτο τρία, κύριε Κρυβό Καπίτσου, παρακαλώ. Όπως προείπα, υπενθυμίζω το θέμα της εμπιστοσύνη. Το πώς έχει τρωθεί η εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία. η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανονικές εκλογές και πάλι και να φανεί στοιχεία στην πολιτική ζωή λόγω της υπόθεσης Atlas. Εδώ με την τροπολογία αυτή υπενθυμίζω την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα Ιδρικά Βαλκάνια ή τις κατάληψης του κράτους και έχουμε και κάποια νούμερα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ναι, όντω υπήρξε απώλεια εμπιστοσύνη γιατί οι εκλογέ αγνοήθηκαν από, την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δυστυχώ αγνοήσει τα αποτελέσματα, θα τα, δεν θα τα είχε αγνοήσει αν είχε κερδίσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την τρία. Ποιο είναι υπέρ, κατά, Τρεις αποχές. Μία. Και τώρα. Μαυροβούνι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οχτώ. Αποχές όχι. Άρα η τρία του κυρίου Κρυβόκαπιτς απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθών Τέσσερα. Από τους πράσινους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ τι προτείνουμε. Ξεχωριστή, μάλλον τα ψηφοφορία. Προσθέτουμε τον όρο αποπολιτικοποίηση και στη συνέχεια καλούμε τον οργανισμό κατά της διαφθοράς να διατηρήσει την ανεξαρτησία του από πολιτικές ε, επιρροές κατά τη διάρκεια της διενέργειας ερευνών για τη διαφθορά. Και τώρα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα με τη λέξη αποπολιτικοποίηση. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας, ε, κατά, τρεις, αποχές όχι. Από το Μευροβούνιο υπέρ, ένας κατά, οχτώ, δεν έχουμε αποχές. Συνεπώς, το πρώτο τμήμα της τέσσερα Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Που καλεί τον οργανισμό κατά της διαφθοράς να δράσει με πνεύμα ανεξαρτησίας χωρίς πολιτικές επιρροές όταν συλλέγει πληροφορίες και διευνά υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων από τους Ευρωπαίους από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4 κατά. Σχολή εκτός μικροφώνου. Συγγνώμη, να του πω στο μικρόφωνο. Χρειάζεται απλώς να διατυπωθεί φράση στον ενεστώτα, όχι στον αόριστο. Α, κοιτάξτε, όλο το κείμενο είναι στον αόριστο. Όλο το κείμενο είναι στον αόριστο, οπότε μην, ε, μην ανησυχείτε. Εντάξει, okay, το κατάλαβα. Λέω και Στάνακ, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Υπέρ, λοιπόν. Κανείς κατά, μηδέν εποχές, άρα το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Και πάμε στην 5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγγνώμη, του κύριου Ράδος. Κατά τμήματα και πάλι, πρώτο τμήμα. Υπάρχει εδώ ένα κείμενο που λέει κάτι υπέρ της αλλαγής της νομοθεσίας. Υπέρ. Τέσσερις. Κατά. Όχι. Αποχές. Όχι. Και τώρα το Μαυροβούνιο. Υπέρ. 9 κατά όχι αποχές 0 άρα το πρώτο τμήμα της 5 του κύριο Ράδος εγκρίνεται δεύτερο τμήμα του κύριο Ράδος και πάλι καλεί τις αρχές να δώσουν αρμοδιότητα στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να αναλύει, να συλλέγει πληροφορίες κλπ. Ευρωβουλευτές υπέρ, ένας κατά, δύο, αποχές, ένας. Μαυροβούνι υπέρ, κατά, οχτώ, αποχή, μία. Οπότε, το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας του κ. Ράδος απορρίπτεται. Τροπολογία 6 του κυρίου Καπίτσου. Έχουμε προτείνωμενη συμβαστική που λέει σημειώνει τη θέση των βουλευτών της αντιπολίτευσης να μην συμμετάσχουν ε, και εδώ σε δύο τμήματα πάμε στο πρώτο τμήμα της συμβαστικής παρακαλώ αυτό που μόλις διάβασα κύριε Καπίτσου θέλετε να εξηγήσετε κάτι εδώ όχι Α, θέλετε το δεύτερο τμήμα να το διαγράψετε, οπότε δεν υπάρχει συμβαστική εδώ. Που λέει καλή όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν μέρο στην μεταρρύθμιση τη εκλογική νομοθεσία κλπ. Αν δεν θέλετε να εξηγήσετε κάτι, κανένα πρόβλημα. Κρυβό καπίτσο. Χαίρομαι που βελτιωνόμαστε. Χαίρομαι που συζητάμε την τεχνική διακυβέρνηση δεν χρειάζεται αυτό να είναι στην ε, συμβαστική. Εν πάση περιπτώσει το ότι αναφέρεται και μόνο εδώ είναι θετικό. Εγώ θα διαβάσω την τροπολογία, λέει πρόεδρο. Α κάνετε την παρατήρησή σα. Λοιπόν, λέει το κείμενο. Θυμίζουμε την απόφαση μελών τη αντιπολίτευση να μην συμμετάσχουν σε καμία μελλοντική απόφαση χωρίς την ε, δημιουργία τακτικής κυβέρνησης. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη συμβαστική. Ποιος είναι υπέρ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερις, κατά, κανείς, δεν έχουμε αποχές. Πολύ ωραία, Μαυροβούνιο υπέρ. Κατά. Όχι εποχές. Δεν εποχή. Α, μία εποχή. Πολύ ωραία. Άρα το πρώτο τμήμα αυτής της τροπολογίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Το πρώτο λοιπόν δεκτό όπως είπα. Δεύτερο. Ευρωβουλευτές υπέρ. Κανείς. Κατά. Τέσσερις. Αποχές. Καμία. Μαυροβούνιοι υπέρ. Μία. Κατά. οχτώ, Αποχές μηδέν. Οπότε το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Και πάμε στην ε, τροπολογία 7 του κυρίου Κρυβόκαπιτς. Εδώ λοιπόν προτείναμε συμβιβαστικές για αποτελεσματική εφαρμογή. Θέλετε να διευκρινίσετε την τροπολογία σας, κύριε Κρυβόκαπιτς. Θα ήθελα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το δεύτερο τμήμα δεν έγινε δεκτό. Εκεί που είναι πιο... Ε, το κομμάτι αυτό είναι πιο σημαντικό. Είναι σημαντικό κομμάτι της μελλοντικής προόδου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε ε, δεκτό. Ευχαριστώ. Είναι συμβιβαστική τροπολογία. Θα διαβάσω για μία ακόμη φορά, λέει ο πρόεδρο. Τονίζεται ακόμα σημασία τη αποτελεσματική υλοποίηση. Ε, Ευρωβουλευτέ, ποιο είναι υπέρ. Τέσσερι εναντίον. Κανένα. Αποχή καμία. Μαυροβούνιο. Ποιο είναι υπέρ αυτή τη τροπολογία. Εννέα. Αποχή καμία. Κανεί κατά. Οπότε συμβαστική αυτή γίνεται δεκτή. Πάμε στην τροπολογία 8. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία από τους ευρωβουλευτές. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 8. 3. Κατά. Αποχές. Καμία. Από το Μαυροβούνιο. Υπέρ. Ένας. Κατά. 8. Αποχές. Καμία. Η τροπολογία 8 δεν γίνεται δεκτή. Πάμε στην τροπολογία 9 του βουλευτού κυρίου κρυβόκαπιτ. Υπέρ από πλευράς ευρωβουλευτών. Ποιος είναι υπέρ της 9. Ένας. Κατά. Τρεις. Αποχές. Καμία. Από τους Μαυροβούνιους ένας είναι υπέρ κατά 8. Αποχές καμία. Η τροπολογία 9 δεν γίνεται δεκτή. Πάμε στην τροπολογία παριθμών 10 του κυρίου Ράντος, του Ευρωβουλευτού. Ποιος είναι υπέρ της 10 τους Ευρωβουλευτές. Τέσσερις. Κάποιος εναντίον όχι, εποχές καμία, από το Μαυροβούνιο Κοινοβούλιο υπέρ του 10, της τροπολογίας 10, 9, καμία αποχή, ουδής εναντίον, οπότε η τροπολογία 10 γίνεται δεκτή. Πάμε στην τροπολογία 11 που υπευλήθη από τους πράσινους την ε, Α, ποιος είναι υπέρ της 11 από τους ευρωβουλευτές, 4. Εναντίον, κανείς, αποχή καμία. Από το Μαυροβούνιο, ποιος είναι υπέρ της 11. 9. Αποχή καμία, ουδέμια ψήφος εναντίον, άρα η τροπολογία 11 των πρασίνων έχει γίνει δεκτή. Τροπολογία 12 του Ευρωβουλευτού κ. Ράντος. Έχουμε προτείνει συμβαστική τροπολογία και λέμε καθώς και καλύτερη, κατα, καλύτερη, πιο αποτελεσματική εκδίκαση στα δικαστήρια των διαφόρων ποινικών αδικημάτων. Ποιο είναι υπέρ, ε, τέσσερι Ευρωβουλευτέ, κανεί κατά, καμία αποχή, υπέρ τη τροπολογία 12, τη συμβαστική μάλλον τροπολογία από πλευρά Μαυροβουνίου, 9 είναι υπέρ της συμβαστικής, εναντίον κανείς, αποχή καμία. Οπότε η τροπολογία αυτή η 9 γίνεται δεκτή, η συμβαστική. Τροπολογία 13 του Ευρωβουλευτού Ράντος. Αυτή η τροπολογία υποδιαιρείται σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Να εξασφαλίσει αποτελεσματική αύξηση των διοργανικών πολιτικών όσον αφορά το φύλλο, τα δικαιώματα των διαμεταφυλικών, ατόμων με αναπηρία, για να διατεθούν αρκετά χρήματα, ούτω ώστε να εφαρμόζονται καλύτερα αυτές οι πολιτικές από τους ευρωβουλευτές. Ποιος είναι υπέρ αυτού του τμήματος. Τέσσερις. Ουδής αναντίον, καμία αποχή από το Μαυροβούνιο υπέρ του πρώτου τμήματος της τροπολογίας. Εννέα. Καμία αποχή, καμία ψήφος εναντίον. Το πρώτο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας γίνεται δεκτό. Το δεύτερο τμήμα. Θέλαμε να διαγράψουμε τις λέξεις όπως γυναίκες, παιδιά, η Ρωμά συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με αναπηρία και ΛΟΑΔΜ. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος του Ευρωβουλευτού. Τέσσερις, καμία ψήφος εναντίον, καμία αποχή από πλευράς Ευρωβουλευτών, από πλευράς Μαυροβουνίων, ποιος είναι υπέρ, εννέα, ουδεμία ψήφο, κατά, καμία αποχή. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας του κυρίου Ράντος γίνεται δεκτό. Το τρίτο τμήμα. Που καταδικάζει το γεγονός ότι έχουμε διεθνωτικά προβλήματα, κάτι που οδηγεί σε ανεπαρκή ε, προστασία των οικογένειών κλπ όταν καθυστερούν οι δίκες όσον αφορά την οικογενειακή βία, ε, καθυστερούν οι δίκες και είναι χαμηλές οι ποινές. Από τους βουλευτές. ποιος είναι υπέρ, τέσσερις, κατά, ε, καμία ψήφος, αποχές καμία. Το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ποιος είναι υπέρ, του τρίτου τμήματος, κανείς, κατά, οκτώ, αποχές καμία. Οπότε το τρίτο τμήμα δεν γίνεται δεκτό. Τροπολογία 14. Κρυβόκαπιτς από το Μαυροβούνιο. Προτείναμε συμβαστική τροπολογία που πάει ως εξή. Τονίζει ότι οι οργανώσεις, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα χωρίς παρεμβάσεις από τους ευρωβουλευτές. Ποιος είναι υπέρ του συμβιβαστικού, οι τέσσερις εναντίον κανείς, αποχές καμία, Μαυροβούνιο υπέρ εννέα. Κατά κανείς, αποχές καμία. Οπότε η συμβιβαστική τροπολογία έχει γίνει δεκτή. Πάμε στην τροπολογία 15 του βουλευτού του κ. Κρυβόκαπιτς από το Μαυροβούνιο οι ευρωβουλευτές ποιος είναι υπέρ? Ότι τα επιτόκια είναι υψηλότερα από το στατιωτικό προπολογισμό. Θέλω να δώσουμε αυτή την εικόνα. Ξέρετε άλλη χώρα στον κόσμο που έχει μεγαλύτερο στατιωτικό προπολογισμό μάλλον ότι δίνει τόσο ψηλά κονδύλια για το στρατό και είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε ουδέτερη χώρα. Ήθελα να δώσουμε την πραγματική εικόνα, τα λένε στοιχεία. Το έλλειμμα του προπολογισμού φέτος είναι 31% μεγαλύτερο από πέρσι. Το πρώτο δεκάμινο του 2018 είχαμε έλλειμμα 38 εκατομμύρια. Τώρα σε αυτούς τους μήνες έχουμε 32 εκατομμύρια. Πέρσι σε 10 μήνες 38. Και θέλαμε να το τονίσουμε αυτό. Για να φανεί η πορεία μας. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ του ευρωβουλευτές, κανείς, κατά. Τρεις, αποχές, μία, δύο. Δύο υπέρ, δύο αποχές. Μαυροβούνιο, υπέρ, μία ψήφος υπέρ, κατά, οκτώ. Αποχές, καμία αποχή. Οπότε τροπολογία 15 Κρυβόκαπιτς δεν γίνεται δεκτή. Ψηφίσουν τροπολογία 16 πρασίνων. Ευρωβουλευτές υπέρ. Θέλετε να εξηγήσετε. Ορίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, την περασμένη φορά ήδη συζητήσαμε τα θέματα τα περιβαλλοντικά και είπαμε καλώς, έχουμε διαφορετικό θέμα σήμερα, α μιλήσουμε για το περιβάλλον την επόμενη φορά. Επίση, πρόκειται περί ανοίγματο του κεφαλαίου 27 και είχατε υποσχεθεί ότι θα συζητήσουμε το περιβάλλον αυτή τη φορά. Το σέβομαι ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν έχετε χρόνο και ότι πρέπει να προχωρούμε. Αλλά εδώ βλέπω στον κατάλογο ψηφοφοριών ότι οι βουλευτές του Μαυροβουνίου θα καταψηφίσουν. Να σα υπενθυμίσω ότι αντιπροσωπεύεται τη χώρα του κόσμου που έχει την οικολογία στο σύνταγμά τη. Η μόνη. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, γεμίστε το με υποσχέσεις και δράση. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που έλεγα, απλώς ε, ε, τα, τα, διάφορα, τα, τα, τις μονάδες υδροπαραγωγικές Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα δύο ποτάμια. Υπάρχουν πολλά προγράμματα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την υδροελεκτρική ενέργεια, αλλά θα πρέπει να δείτε ότι κινδυνεύεται μακροπρόθεσμη ευημερία και εισόδημα μέσω τουρισμού που μπορείτε να αναπτύξετε σε αυτούς τους πολύτιμους ποταμούς, τη πλούσια φυσική σας κληρονομιά. Κάντε θυσίες για βραχυπρόθεσμο κέρδος που μόνο μία εταιρεία παραγωγής τεχνικής ενέργειας έχει σαν εισόδημα. Ανταυτού μπορείτε να έχετε μακροπρόθεσμο εισόδημα, ανάπτυξη τυπέθρου πέθρου για όλη την περιοχή, ευημερία που θα διαδοθεί στον ντόπιο πληθυσμό και δεν θα τα μαζεύει όλα μία απλή εταιρεία που χρησιμοποιεί τα ποτάμια. Είναι η πιο πολύτιμη φυσική κληρονομιά που έχετε. Ξανασκεφτείτε την αποφασή σας που λέτε ότι δεν είσαστε υπέρ ή να προτείνουμε μια τροπολογία συμβαστική, αλλά κατά ψήφιση νομίζω ότι είναι πολύ απογοητευτικό. Ευχαριστώ κύριε Βάης. Να σας πω ότι είναι μονοήμερη συζήτηση της Επιτροπής αυτής και έγινε κατόπιν αιτήματο των Ευρωβουλευτών. Δεν συντομεύσαμε εμεί τη διάρκεια τη συζητήσεω. Εμεί είμαστε ανοιχτοί να συζητούμε αυτά τα θέματα. Εσεί ζητήσατε να είναι μόνο ημέρα. Συμφίσουμε την τροπολογία των Πρασίνων και τη Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Ευρωβουλευτών. Ποιο υποστηρίζει την ε, τροπολογία αυτή. Δύο. Κατά. Μία ψήφο. Αποχέ. Μία. Από το Μαυροβούνιο υπέρ ένας. Κατά οκτώ Αποχές καμία. Άρα αυτή η τροπολογία δεν ενεκρίθη. Ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τροπολογία 17. Ράντος. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 17. Ευρωβουλευτές 4. Κατά. Ουδής. Καμία αποχή. Ποιος είναι υπέρ από το Μαυροβούνιο. 9. Κατά. Ουδής καμία αποχή. Οπότε θεωρούμε ότι η τροπολογία ράντος ενεκρίθη. Εγκρίνεται. Τώρα για την τελική ψηφοφορία του σχεδίου συστάσεων. Οι ευρωβουλευτές να ψηφίσουν. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Τρεις. Κατά. Μία ψήφος. Αποχές. Καμία. Από το Μαυροβούνιο οι βουλευτές. Υπέρ του σχεδίου συστάσεων με τις τροπολογίες που έγιναν 8. Κατά μία ψήφος. Αποχές καμία. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε εγκρίνει το σχέδιο αυτό των συστάσεων το σχέδιο δήλωσης στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Έχει κάποιος θέμα για, τα... για αυτό το σημείο. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Σημείο 8. Τόπος και χρόνος της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής. Η επόμενη συνεδρίαση Α, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα πρέπει να γίνει τον Οκτώβριο του 2019 στην Ποντγκορίτσα. Πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, να ευχαριστήσω τον συμπρόεδρο, τον κύριο Μάρτιν και την αντιπροσωπεία του και τον κύριο Χακ Λάιτερ, τον συνάδελφο. Ευχαριστώ τη γραμματεία για τη βοήθεια Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, τη 17η συνεδρίαση της Επιτροπής μας, η οποία ολοκληρώθηκε. Γεια σας. Καλό βράδυ.